Και τώρα, επόμενο θέμα στην στη διάταξη. Το Διοικητικό Δικαστήριο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητων. Και δίνω το λόγο στον κύριο, στον πρόεδρο, προεδρεύοντα Λεσκεβίτσιους. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κύριε Επίτροπε, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ε, είναι ένας διεθνής ε, θεσμός, μόλον ότι αυτοί που έχουν βάλει την υπογραφή τους είναι 17 οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμός είναι ένα ξεχωριστό φορέα και δεν αποτελεί μέρο του νομικού πλαισίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο, συνεπώς, δεν είναι αρμόδιο για να συζητήσει θέματα που αφορούν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό και δεν έχει συζητήσει το θέμα της δημιουργίας ενός διοικητικού δικαστηρίου για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Πέραν αυτού, επειδή η Λιθουανία δεν ανοίγει στο Μηχανισμό Σταθερότητας, δεν μπορεί να εξετάσει αυτό το θέμα ως μέλος του μηχανισμού. Ο ίδιος ο, ο μηχανισμός θα μπορούσε να απαντήσει καλύτερα στα ερωτήματά σας. Θα ήθελα να πω ότι εγώ καταλαβαίνω ότι το άρθρο 23 που εγκαθιδρύει το μηχανισμό που συνεπάγεται και την υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει τις συνθήκες που αφορούν την πρόσληψη του ε, Διευθυντή αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία. Πέρα από αυτή τη διάταξη, το άρθρο 18 αναφέρει ότι η κανόνες θα πρέπει να καθορίζουν τις διαδικασίες σε ό,τι αφορά διαμαρτυρίες που προέρχονται από τις χώρες μέλη. Συνεπώς, τα μέτρα αυτά αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου δικαστηρίου από τα σχολεία μου νομίζω ότι θα κατανοήσετε ότι δεν είμαι σε θέση να κρίνω την καταλληλότητα ή το σκόπιμο της δημιουργίας αυτού του δικαστηρίου. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι είναι σημαντικό από την άποψη της διακυβέρνησης να, μπορεί, να μπορούν να, εξεταστούν θέματα από έναν ανεξάρτητο φορέα. Παρεφερεί δικαστήρια υπάρχουν σε άλλα διεθνή θεσμικά όργανα όπως για παράδειγμα την Παγκόσμια Τράπεζα ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καταλαβαίνω ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για να περιστούν τα προβλήματα που αφορούν τη δημιουργία αυτού του διοικητικού δικαστηρίου. Τα μέλη θα αμείβονται για κάθε συνάντηση και δεν θα λαμβάνουν κάποιο ε, μηνιαμισθό. Τα θέματα τα, οι δεν αποκλείουν τα μέλη αυτά από οποιαδήποτε άλλη ε, από οποιοδήποτε άλλο φορέα με, ε, πέρα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ε, Σταθερότητα. Και δεν θα επηρεάσει αυτό το προπολογισμό τη κοινότητα. Σε ό,τι αφορά το προπολογισμό του Μηχανισμού Σταθερότητα, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τους, ίδιο, τον ίδιο το φορέα. Αξιότιμα μέλη, είμαι σίγουρος ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Μηχανισμού έχει ζυγίσει τα πλεονεκτήματα τη δημιουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου. Το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού δεν είναι η υπάλληλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οποιαδήποτε απόβαση να δοθεί αυτός ο ρόλος θα μπορούσε να επηρεάσει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σας είπα, καταρχάς, αυτό δεν είναι ένα θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου. Θα έλεγα ότι θα ήταν σκόπιμο να απευθυνθείτε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και στους φορείς που τον διοικούν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως είμαστε πολύ περίεργοι. Δεν ξέρω να δούμε τι θα πει η Επιτροπή. Και δίνω τον λόγο στον Αντιπρόεδρο κ. Σεύκοβος και πάλι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, αγαπητέ Υπουργέ. Θέλω να αρχίσω με ευχαριστίες προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ερώτηση, γιατί δείχνει ότι όλοι ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για την ανάπτυξη παρετέρω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που έχουμε για να δώσουμε απαντήσεις στην κρίση και από αυτόν εξαρτάται η συνέχεια που θα δοθεί και η απάντηση που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συνεχίζει να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη σταθερότητα και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και θα το κάνει αυτό και στο μέλλον. Η Επιτροπή λοιπόν στηρίζει απόλυτα όλα τα μέτρα που θα διασφαλίσουν τις βέλτιστες πρακτικές όσο γίνεται περισσότερο και σε αυτό το μηχανισμό. Για το θέμα που μας απασχολεί σήμερα πρέπει να υπογραμμίσουμε αυτό που λένε και στην ερώτησή τους ε, οι ευρωβουλευτές, ότι πρόκειται για ένα ανεξάρτητο όργανο εκτός συνθήκων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παρατηρητής μόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο και συμβάλλει με τις γνώσεις της. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός ε, Σταθερότητας έχει περίπου 100 άτομα προσωπικό. Πρέπει να υπάρχει ελαστικότητα για να προσαρμόζεται στις διάφορες καταστάσεις. Αυτό έχει να κάνει με την απασχόληση και στη συγκεκριμένη περίπτωση και με τα θέματα προσφυγών των υπαλλήλων. Το δικαστήριο θα έπρεπε να επιτρέπει τους υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Μηχανισμού Σταθερότητας να προσφεύγουν για αποζημιώσεις ή για οτιδήποτε άλλο. Όπως συμβαίνει και με άλλα οικονομικά ιστιτούτα, όπου είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, το Εθνικό Μεσονατικό ε, Ταμείο κλπ. που έχουν αντίστοιχα διοικητικά δικαστήρια το καταστατικό και ο κανονισμός γενικότερα έχουν ήδη εγκριθεί από το Δικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και τους εκπροσώπους όλων των πλευρών. Σύμφωνα με την διοικητική δομή και με τις ευθύνε έτσι όπως αυτές αναφέρονται στην συνθήκη ιδρυσής του. Θα σταθώ όμω ε, εδώ λίγο για να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Πρώτον, το Δικητικό Δικαστήριο θα αποτελείται από πέντε ανεξάρτητα μέλη που θα κρίνουν τις προσφυγές και άλλα διοικητικά θέματα. Τα άτομα αυτά δεν θα μπορούν να καταλαμβάνουν άλλη θέση ούτε πριν, ούτε κατά τη διάρκεια, ούτε μετά τις θητείες τους αυτή στο Διοικητικό Δικαστήριο στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας δεν θα μπορούν να έχουν άλλο πόστο. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό. Το κόστος τώρα το οποίο έχει να κάνει με τα άτομα αυτά θα το υπομειστεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και θα εξαρτηθεί από τις υποθέσεις που θα επεξεργάζονται και δεν θα έχουν καμία μόνιμη θέση. Η αμοιβή αυτή είναι απόρριτη. Όμως η δομή θα αντιστοιχεί στην δομή αμοιβών που έχουν δικαστές σε άλλα διεθνή όργανα. Τέλος, τα άτομα αυτά, όπως σας είπα, δεν θα μπορούν να έχουν καμία θέση απολύτως στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας άλλη. Τώρα δεν υπάρχει καμία πρόθεση να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό και ούτε πρόκειται να υπάρξει κατάχρηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού σταθερότητα. Δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις στον κοινοτικό προπολογισμό. Έτσι έρχομαι στην πρώτη επιμέρους ερώτηση που λέει γιατί είναι εφικτό ένα διοικητικό δικαστήριο. Το άρθρο 3 της Εθήκης λέει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσώπων όλων των μερών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού σταθερότητα. θα αποφασίζουν για τις ειδικές κάτω από τις οποίες θα προσλαμβάνεται προσωπικό. Υπάρχει καταστατικό για το προσωπικό που αναφέρεται στα δικαιώματα του προσωπικού, στις συνθήκες πρόσληψης και αναφέρει και τη δημιουργία του διοικητικού αυτού δικαστηρίου. Όλα τα έγγραφα αυτά πρέπει κανείς να τα διαβάσει βέβαια στο σύνολό τους. Και κάτι ακόμα. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας προσπάθησε να εξετάσει και την ανελακτική που προτείνουν οι ευρωβουλευτέ. Δηλαδή, μήπω θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το Ευρωπαϊκό, Δικαστικό, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τι περιπτώσει αυτέ. Αλλά δεν είναι τόσο απλό το θέμα όσο ίσω φαίνεται εκ πρώτη άψεω. Διότι ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα δεν είναι ευρωπαϊκό όργανο ή υπηρεσία και γι' αυτό δεν έχει απευθεία πρόσβαση στην νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Οπότε, προκειμένου ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα και το προσωπικό να μπορεί να έχει πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, προηγουμένω πρέπει να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο βέβαια θα πάρει χρόνο, 18 μήνε περίπου. Και μια που υπάρχουν ε, πολλέ ε, πλευρέ, δεν μπορεί να γίνει μονομερός ούτε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ούτε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητα. Και δεν είναι κάτι που μπορεί να λυθεί εύκολα και γρήγορα. Στο μεταξύ, ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα πρέπει να αποφασίσει πώ θα προχωρήσει. Δεν μπορεί να αγνοήσει την ανάγκη να υπάρχει ένα δικαστήριο που θα επιλύει προσφυγές των υπαλλήλων. Συνεπώς, δημιουργείται το διοικητικό δικαστήριο στο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα να συμμορφώνεται πλήρω με τι βέλτιστε πρακτικέ και να μπορεί να επιλύει θέματα προσωπικού. Και κάτι τελευταίο πριν σας δώσω σε εσά το λόγο και πάλι. Να ξέρετε ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας προσπάθησε να βρει την κατάλληλη απάντηση. Ξεκολουθεί να είναι ένα όργανο με διοικητικές διαδικασίες που θέλει να τηρεί τους κανόνες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ τους συναδέλφους να λάβουν υπόψη στο τέλο τη συζητήσεως. Δεν θα έχουμε περιθώριο για ε, διαδικασία κάτω στη ΆΗ, ούτε και για μπλε κάρτε. Θα ακούσουμε όμω τώρα τον κύριο Έλμαρ Μπρόκ, εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, είμαι συγκλονισμένος από τον τρόπο ένα θέμα τόσο σημαντικό για την κοινοτική πολιτική, για το ευρώ είναι κοινοτική πολιτική, ε, τοποθετούνται το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Είμαι συγκλονισμένο ιδιαίτερα στον τρόπο που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί από το Συμβούλιο το περίμενα σχεδόν. Και θα ήθελα ασφαλώς να αναφερθώ στις παρατηρήσεις του κυρίου Σεύκοβιτς ότι είναι πιθανή η χρήση του ευρωπαϊκού σε δικασίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μας λέτε είναι πιθανόν, είναι δυνατόν. Δεν δίνεται απαντήσει όμως στα ερωτηματικά μας. Γιατί το να υπάρχει για 100 άτομα προσωπικό ένα διοικητικό δικαστήριο, ανεξάρτητο της σημασίας του έργου του, είναι γελίο καταρχάς. Δεύτερον, ο ευρωπαϊκός αυτός ε, μηχανισμός σταθερότητας για τον οποίο άνοιξε ουσιαστικά ο δρόμος για συμμετοχή και παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί είναι μηχανισμός της Ένωσης και έχουμε κάνει εμείς ε, σχετική έκθεση. Το να συνδυάζεται με ένα τέτοιο ειδικό δικαστήριο επίσης δεν έχει κανένα νόημα. Αποτελεί για ένα πολύ σοβαρό πλήγμα στα ευρωπαϊκά όργανα και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και βέβαια την ενότητα της νομολογίας που θα προκύψει από δύο διαφορετικά δικαιοδοτικά όργανα. Και ξεκάθαρα μια αποτελεί μια επιλογή εσφαλμένη, ένα δρόμο λάθος που απορώ πως είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς ουδεμία ε, ουδένα ερωτηματικό, χωρίς ουδένα προβληματισμό να ακολουθεί τον δρόμο αυτόν. Ούτως ή άλλως και για τον προϋπολογισμό τον ευρωπαϊκό θα ήταν πολύ πιο απλό να, ήταν, να, είχε, να υπαγόταν αυτή η διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να μην χρειάζεται κάποιοι δικαστές του ειδικού του διοικητικού αυτού δικαστηρίου για τα 100 συγκεκριμένα άτομα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σταθερότητα να ασχολούνται με κάποιε υποθέσει. Για να μην μιλήσουμε, κύριε Προεδρεύων, για Παγκόσμια Τράπεζα και άλλα όργανα. Το να μα λέτε ότι κάπου στη Ουάσιγκτον υπάρχει ένα όργανο το οποίο έχει αντίστοιχου ε, ε, αντίστοιχου μηχανισμού δικαιοδοσία είναι γελίο και αποτελεί βέβαια απόδειξη έλλειψης πολιτικής βούληση, έλλειψης πολιτικού ορώματο και μόνο το γεγονό ότι θέλετε να έχετε ένα όργανο το οποίο αρχίζει να λειτουργεί και μετά με αρχίσει να λειτουργεί λέτε Αχ, να κοιτάξουμε να δούμε εάν χρειάζεται παραπάνω κάτι να του συμπληρώσουμε γιατί αυτό οδηγεί βέβαια σε κατακαιρματισμό τη Ένωση και τη πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί μιλούμε για μια πολιτική τη Ένωση, γι' αυτό θεσπίστηκε το όργανο αυτό και δυστυχώς υποσκάπτεται η πολιτική της Ένωσης διαρκώς όλο και περισσότερο. Όπως είπα αισθάνομαι συγκλονισμένος και δεν μπορούσα παρά να εκφράσω τη θλίψη μου, ιδιαίτερα για τις τάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκουαλτιέρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να πω ότι και εγώ δεν είμαι πουδενή ικανοποιημένος με τις απαντήσεις που έδωσε το Συμβούλιο και η Επιτροπή στα ερωτήματά μας. Δίχως άλλο, το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας είναι μια διακυβερνητική οργάνωση, το γνωρίζουμε καλά. Εάν θέλουμε όμως να ακολουθήσουμε αυτή την οδό και να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία σχέση με αυτό, δεν καταλαβαίνω γιατί το Συμβούλιο και η Επιτροπή επισήλθαν σε λεπτομέρειες, μας εξήγησαν ε, το το ένα άρθρο, το άλλο ε, άρθρο γιατί ποιε ήταν οι επιπτώσει στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ότι θα χρειαστούν 18 μήνε κτλ. κτλ. Αν δεν έχει καμία σχέση, η μοναδική λογική απάντηση θα ήταν να μην απαντήσουμε. Επειδή έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το ξέρουμε καλά γιατί βασίζεται στην Επιτροπή και οι αποφάσεις περνάνε από το Eurogroup και υπάρχει και σε ένα άρθρο της συνθήκης το οποίο τροποποιήσαμε. Είναι απόλυτα ξεκάθαρο ε, Μάλλον θα έλεγα ότι είναι γελίο να πούμε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τον μηχανισμό σταθερότητας. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξεφύγουμε από ένα πρώτο βασικό ερώτημα. Πώς συμβαίνει το διοικητικό δικαστήριο να καλύπτει 50.000 άτομα με 7 δικαστές και για την ίδια δουλειά χρειάζονται 5 δικαστές για 100 άτομα. Αυτή είναι μια λογική χρήση των χρημάτων ε, των ε, φορολογούμενων και ποιος ασκεί τον έλεγχο. Το Κοινοβούλιο όχι, δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Εθνικά Κοινοβούλια μπορούν να το κάνουν. Τι είναι αυτός ο μηχανισμός γίνεται, αρχίζει να είναι κάτι που τίθεται εκτός ελέγχου. Και αυτό το μικρό επεισόδιο που δεν είναι και τόσο μικρό, είναι ένα ανησυχητικό σύμπτωμα μιας τάσης που ε, όταν ε, εμείς εκφέραμε άποψη για την τροποποίηση του 136 είπαμε ότι ε, υπήρξε μία ένδειξη και στο, στην απόφαση του Συμβουλίου. Ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε αφορά την ολοκλήρωση των, ε, του μηχανισμού σταθερότητας. Ε, μία ενσωμάτωση και όχι μία απομάκρυνση. Ο κύριος Εύκοβης είπε ότι πραγματικά το Διοικητικό Συμβούλιο εξήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματικά είναι ακατανόητη η επιλογή των κρατών μελών να εξουσιοδοτήσουν αυτό τον οργανισμό να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και θα πρέπει να πω με μου ότι είναι πραγματικά γελία η αιτιολόγηση του εκπροσώπου του Συμβουλίου σύμφωνα με τον οποίο πέντε δικαστές για 100 άτομα είναι οικονομία. Ενώ όταν χρησιμοποιήσουμε τους επτά δικαστές που καλύπτουν 50.000 θα είχε ένα ε, κόστος ε, για τον ευρωπαϊκό ε, προϋπολογισμό. Γιατί όλα τα μέλη τα Ένωση είναι μέλη του μηχανισμού, όλα τα μέλη της, του μηχανισμού είναι και μέλη τη ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώ, θα ήθελα να το πω με σαφήνεια ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα σταματήσει να ελέγχει τον μηχανισμό σταθερότητας και θα καλέσει τις χώρες μέλη μέσω της συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια να απαντήσουν για μια πολιτική επιλογή που αποτελεί ανησυχητική ένδειξη ότι παίρνουμε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θα έπρεπε να παίρνει η διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκίγκολ. Κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς πρέπει να εκφράσω την έκπληξή μου για τη δικασία αυτή. Για 100 εργαζόμενους, ένα διοικητικό δικαστήριο 5 μελών για τα διοικητικά θέματα. Ενώ υπάρχει ευρωπαϊκό δικαστήριο με ειδικό τμήμα για τα εργασιακά ζητήματα. Οι απαντήσεις δεν που μας δίνετε στις ερωτήσεις μας, γιατί θεωρείται απαραίτητο αυτό, τι είδου ε, χρήση μπορεί να έχει μέσα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα και γιατί πρέπει να αναπτυχθεί έτσι ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα, το Συμβούλιο μα λέει: Α, κοιτάξτε, ρωτήστε το, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα. Αυτό όμω έρχεται σε απόλυτη αντίθεση και αντίφαση με αυτά που μα είχε πει με το, ε, το Συμβούλιο όταν θεσπίστηκε στι 25 ε, Μαρτίου του 2001, λέει ο μιλητή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου είπατε, υποσχεθήκατε πως το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώνουν τακτικά για τις διαδικασίες, για τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Είχατε αναλάβει δηλαδή τη σχετική ευθύνη να δίνετε απαντήσεις σε μας τώρα, να μας παραπέμπετε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, σημαίνει ότι δεν τιμάτε τις δεσμεύσεις της εποχής εκείνης. Και ε, έχοντας το μεταξύ μετατρέ... έχετε το μεταξύ μετατρέψει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητα ε, σε διακυβερνητικό όργανο στις 25 Σεπτεμβρίου του 2013 κάλεσαμε τον κύριο Ρίκλινγκ να έρθει να μας μιλήσει αλλά αρνήθηκε συγκεκριμένες ερωτήσεις να τις απαντήσει απαντήσεις που είχαν να κάνουν με τη λειτουργία του μηχανισμού και ιδιαίτερα με την Ευρωζώνη και έτσι ήταν σαν να κυνηγάει ο σκυλό στην ουρά του. Το ένα γύρναγε γύρω πίσω από το άλλο. Δεν δόθηκαν απαντήσεις και γι' αυτό θέλω να σα ρωτήσω πόσο τάσεστε εσεί προς τη δημιουργία ενός νέου δικαιοδοτικού οργάνου και θέλω την, από την Επιτροπή γραπτά να μου εξηγήσει ποια νομοθεσία, με ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για να ε, για να ε, προσκοληθεί το δικαστήριο αυτό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ώστε να εξοικονομηθούν κονδύλια προς όφελος των Ευρωπαίων φορολογουμένων γιατί δεν χρειάζεται και άλλο γραφειοκρατικό όργανο με διακυβερνητικές διαδικασίες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ κύριε Γίγκολτ. Άλλους ομιλητές δεν έχουμε. Ο κύριο Σεύκοβιτ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούω ότι συζητιέται πως το όργανο αυτό φτιάχτηκε με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό πρέπει πάντα να διασφαλίζεται ότι κάθε βήμα γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και με τις βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης όπως σε αντίστοιχα δημοσιονομικά ιδρύματα. Από αυτή την άποψη λοιπόν αντιλαμβάνομαι γιατί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θέλησε να φτιάξει διοικητικό δικαστήριο, γιατί αυτή είναι η βέλτιστη πρακτική. Ήταν αυτό που έλειπε για να μπορεί να εξετάσει προσφυγές των ε, υπαλλήλων ή άλλες διαφορές που μπορεί να υπήρχαν με τους υπαλλήλους του. Συγχρόνως βέβαια, συμφωνώ μαζί σας για το ότι αν συγκρίνουμε το έργο του Διοικητικού Δικαστηρίου και με τον αριθμό των υπαλλήλων που έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που δεν καλύπτει 100 αλλά πάνω από χιλιάδες υπαλλήλους, αντιλαμβάνομαι ότι η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Και ότι θα μπορούσε, όπως λέτε, να καλύψει και τους 100 αυτούς υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Λέτε ότι αυτή θα ήταν η καλύτερη λύση. Ναι, χρειάζεται όμως χρόνος για να γίνει αυτό. και εφόσον μάλιστα δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στον προπολογισμό, είναι κάτι που πρέπει να το αναφέρουμε. Πάντως, ως μόνιμη λύση θα έπρεπε να προτείνουμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας να αρχίσει προπαρασκευαστικό έργο για να δει μήπως τελικά οι προσφυγές των υπαλλήλων θα μπορούσαν να καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στη συνέχεια. Μία δυνατότητα υπάρχει. Η δυνατότητα αυτή είναι να υπογραφεί συμφωνία ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να σας δώσουμε λεπτομέρειες για νομικές απαιτήσει για μια τέτοια συμφωνία. Πάντως από την ανάλυση που έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι μια διαδικασία όπως σας είπα και πριν η οποία θα κρατήσει κάπου 18 μήνες. Συνεπώς όλα θα εξαρτηθούν από την απόφαση που θα πάρουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Σε αυτό η Επιτροπή είναι μόνο παρατηρητής. Εκείνοι θα αποφασίσουν αν θέλουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο ή όχι. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Και τώρα παρακαλώ. Το κύριο Μπρόκ να μην στήσει για το λόγο. Ε, θα δώσω το λόγο στο Συμβούλιο. Mr. President, uh, honorable Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όλες οι παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας θα αναφερθούν στους συναδέλφους μου. Φαίνεται ότι η απόφαση δημιουργίας του μηχανισμού σταθερότητας παρέχει κάποια προστασία στα, ε, στους εργαζόμενους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στα... Για διεθνείς οργανισμούς χρειάζονται άλλες λύσεις. Ε, αυτή είναι μια απόφαση που λήφθη από τους φορείς που διοικούν τον μηχανισμό σταθερότητας. Δεν έχει αποκλειστεί όμως η δυνατότητα να υπάρξει προσφυγή στο, να στραφούν προς το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τι όμως είναι μια απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί από τους ηθήνοντες του μηχανισμού. Είμαι σίγουρος ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες πριν αποφασίσουν, πριν πάρουν τις αποφάσεις τους. Έχω τη βεβαιότητα ότι ο μηχανισμός σταθερότητας γνωρίζει τις απόψεις που εξέφρασαν εδώ τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Από ό,τι φαίνεται ότι είναι η τελευταία φορά που παρίσταμε εδώ, εξ του Συμβουλίου, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία αυτή για να σας ευχαριστήσω όλους για την υπομονή σας, να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής και να σας ευχαριστήσω και για την συνεργασία σας κατά τη διάρκεια της Λιθωνικής Προεδρίας. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ. Μπορεί να ακούστηκαν επικρίσεις. Πιστεύουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντως ότι η Λιθουανική Προεδρία ήταν πολύ δραστήρια στη συμμετοχή της στις συζητήσεις, ήταν πολύ συχνά παρούσα και την ευχαριστούμε. Και τώρα ολοκληρώνεται τη συζήτηση και ελπίζω ότι κατά την εκλογική περίοδο δεν θα έχουμε να συζητήσουμε το μηχανισμό σταθερότητας. Είναι αρκετά περίπλοκη η δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν χρειάζεται να